we open the meeting, uh, can we adopt the draft agenda with the following modification? Uh, να ξεκινήσουμε μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη στο 15 ε, αστική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα σήμερα λόγω του ότι ο εισηγητής απουσιάζει και η ανταλλαγή απόψεων θα αντικατασταθεί με μια σύντομη ανακοκκίνωση που θα γίνει σήμερα γύρω στις 12 με 12.30. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις γλώσσες εκτός από κροατικά και καλωσορίζουμε ένα νέο μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, τον κύριο Άμιαντ Μπασίρ. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εδώ, είναι νέο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας, εκ μέρους της ομάδας ECR, τον καλωσορίζουμε. Επισκέπτες θα έχουμε μία ομάδα σήμερα το απόγευμα, προσκεκλημένων, της, ε, ενός μέλους της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης για τις ε, για το TTIP, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και αν εξέχασα να πω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 21ης και της 22ης Ιανουαρίου 2015, ναι, και τώρα θα περάσουμε στις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Η πλήρης ανταλλαγή απόψεων για το προσχέδιο θα γίνει στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 5 Μαρτίου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου 2015 στις 12 το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι εδώ η Μαριάν Χάρκιν. Γιατί θα σας δώσω το λόγο τώρα ως εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα σα μιλήσω γιατί δεν μιλάμε. Δεν έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Το σχέδιο γνωμοδότηση διανεμήθηκε στου Κιώδη την προηγούμενη εβδομάδα και διατέθηκε και στα μέλη. Σήμερα το πρωί έγινε ε, συζήτηση στην ε, έκτακτη συνεδρίαση στι 5 ε, ε, στις 5 Μαΐου θα γίνει η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων. Ξέρω ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλά μέλη, αλλά δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό. 1500 λέξεις είναι όλη και όλη η γνωμοδότηση και θα γίνει η πλήρης ανταλλαγή απόψεων την επόμενη πέμπτη το πρωί στο μεσοδιάστημα βεβαίω είμαι διαθέσιμη για κάθε μέλος να συζητήσουμε αν θέλει έχουμε λίγο χρόνο αλλά ε, προσβλέπω σε πολλές τροπολιποιήσεις και σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Πολύ οι εισηγητές είναι εδώ στην αίθουσα. Υπάρχει κάποιος που σας θα ήθελε να πει κάτι για το θέμα αυτό. Όχι. Θα το ξανασυζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μα. Θέλει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει κάτι σε αυτή τη φάση. Όχι. Οπότε το αφήνουμε για τώρα το θέμα αυτό. Και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, μέσα ατομικής προστασίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης και θα δώσω τον λόγο στη Λάουρα Άγγια, την εισηγήτρια, τη συντάκτρια της, ε, του σχεδίου γνώματος. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Να πω καταρχήν ότι ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δόθηκε ε, να επιλεγώ ως εισηγήτρια για αυτή την ε, γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη που εκ των προτέρων ε, τοποθετήσατε σε μια εκπρόσωπο ομάδας που, μιας ομάδας που δεν ε, συγκεντρώνει πάντα θετικά βλέμματα να πω ότι προσπάθησα στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης να κινηθώ προς δύο βασικές ε, κατευθύνσεις τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές σε αυτή την υπόθεση. Η οδηγία η οποία θα αντικατασταθεί από αυτόν τον κανονισμό είχε κατά τη γνώμη, περιείχε ε, κατά τη γνώμη μου κάποιες ελλείψεις. Εργαζόμενοι και προσπαθώντας να προετοιμάσω τροπολογίες ε, με βασικό στόχο και προτεραιότητα να καταστεί η προηγούμενη οδηγία ένα υλικό το οποίο να μην δίνει λαβή για ερμηνείες ε, διάφορες, κυρίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. έτσι ώστε να αποφύγουμε διάφορες, ε, πολλές και διάφορες ερμηνείες που θα αποδυναμώσουν την αποτελεσματικότητά της. Πιστεύω πως ε, είναι πολύ σημαντική η ατομική προστασία για την πρόληψη των συχνά θανάσιμων ατυχημάτων, εργασιακών ατυχημάτων. Ε, δώσα λοιπόν μεγάλη σημασία σε αυτό που έπρεπε να θεωρηθεί ως ασφάλεια ε, για τα μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους που τα χρησιμοποιούν και ε, τους οποίους προστατεύουν. Αυτό που προσπάθησα να επιτύχω μέσω των τροπολογιών που υπέβαλα ήταν ότι μόνο χρησιμοποιώντας ε, ε, μέσα ad hoc με διάφορες προδιαγραφές μπορεί να είναι εγγυημένη η ασφάλεια τη στιγμή της εργασίας τους. Και γι' αυτό προσπάθησα να διαφοροποιήσω τη διάφορα μέσα ώστε να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά τα σωματικά των ανδρών, γυναικών, των νέων εργαζόμενων ή των ατόμων με ειδικέ ανάγκε ή με κάποια αναπηρία. Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, στην Ιταλία, αλλά πιστεύω και σε άλλε χώρε τη Ένωση, η οικονομική κρίση καθόρισε, για παράδειγμα, την είσοδο στην αγορά εργασία νέων εργαζομένων που χρειάζεται λοιπόν να φέρουν μέσα ατομική προστασίας προσαρμοσμένα στη σωματική τους κατατομή για να μπορούν να εγγυηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ασφάλειά τους. Επέτυχα, ε, μάλλον θεώρησα ότι έπρεπε να υπογραμμιστεί επίσης η κατάλληλη ενημέρωση και γνώση για το ποιος παράγει ε, κάθε φορά τα μέσα ατομική προστασίας, ποιο τα χρησιμοποιεί και ποιο τα φοράει. Ε, γι' αυτό και πρότεινα μια τροπολογία που προωθεί στην ενημέρωση και στην επικοινωνία ακόμα και εκεί όπου συχνά είναι δύσκολο να διεισδύσει, να χρησιμοποιηθούν και μέσα όπως εφαρμογές ή το, η διάφορα site του ίντερνετ που ε, καθιστούν την ενημέρωση ε, προσιτή. Η ενημέρωση η οποία θα πρέπει να είναι σαφής και γι' αυτό και ζήτησα η ετικέτα τοθεσία η σήμανση για αυτά τα μέσα να υπογραμμίζεται στη γλώσσα της χώρας που τα διαθέτει στην αγορά. Προτείνω ελέγχους και επαληθεύσεις όσον αφορά την πρακτική χρήση και την συμμόρφωση των προϊόντων αυτών με συγκεκριμένους κανόνες. Γιατί μόνο μέσω συγκεκριμένων ε, ελέγχων θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ε, ορθή χρήση αυτών των μέσων. Επίσης ο έλεγχος θα πρέπει να ε, τονίζει που υπάρχει παραβίαση του νέου κανονισμού. Οι κυρώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν μια παράμετρο που θα οθήσει τα κρατημέλη που υιοθετούν και που ε, ακολουθούν αυτό τον κανονισμό να προβαίνουν σε επαληθεύσεις, σε ελέγχους έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται στην αγορά με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, πέρα από αυτό... Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να γίνεται και μία ε, ε, παρακολούθηση ε, κεντρικού τύπου από πλευράς των κρατών και της Κομισιόν με ενημέρωση δικτύου, δικτυωμένη με τρόπο ώστε οι σωστές πρακτικές να αποτελούν κίνητρο για τις διάφορες χώρες που εφαρμόζουν τον κανονισμό. Προσπάθησα πραγματικά να σκεφτώ τους εργαζόμενους, να σκεφτώ όσους κατασκευάζουν αυτά τα μέσα προστασίας, έτσι ώστε πραγματικά να προστατευτεί η ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί μόνο μέσω αποτελεσματικών μέσων και σωστής ενημέρωσης, μόνο ε, μέσω σωστών και αποτελεσματικών ελέγχων μπορούμε να εγγυηθούμε ε, την, την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να συνομιλήσω με οποιονδήποτε θέλει να συνεργαστεί ή έχει περαιτέρω ενδείξεις ώστε να κάνουμε μια ομαδική εργασία και που θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία που θα έχει αυτός ο κανονισμός για την ασφάλεια της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Είμαι λοιπόν ανοιχτή σε διάλογο επικοδομητικό και που να λαμβάνει υπόψη πραγματικά αυτούς που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για να ε, προστατεύσουμε την υγεία τους και την ασφάλειά τους. Σας ευχαριστώ. Ε, thank ε, Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης ηγητές που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Κράσος από το ΕΛΚ. Ε, Cari grazie, buongiorno. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, καλημέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη Λάουρα ε, για την εργασία που έκανε σε αυτό το θέμα. Το να υπάρχουν μέσα ατομικής προστασίας υψηλού επίπεδου μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι σαφές ότι εφόσον μιλάμε για για αυτό το είδος της θέσης απασχόλησης ε, υψηλού κινδύνου το να υπάρχει ας πούμε ένα σωστό μέσο ατομικής προστασίας το οποίο λειτουργεί ορθά αυτό μπορεί να σημάνει τη διαφορά για την ασφάλεια της υγείας του εργαζομένου. Πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί όντως να φέρει ωφέλη σε, ε, από την εναρμόνιση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, γι' αυτό και συμφωνώ με την αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας από έναν κανονισμό. Το εντοσχέ που έχουμε, το φάκελος που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα, ε, παριθμίζει διάφορα καλά σημεία ώστε να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν. Και συγκεκριμένα, προσωπική προσαρμογή για τον τελικό χρήστη για αυτά τα μέσα, ανάλογα με το αν αυτός ο χρήστης είναι άντρας, γυναίκα, νέος ή άνθρωπος με ε, ειδικέ ανάγκες. Έπειτα, ε, εφαρμογή για το smartphone που ε, θα δίνει ε, πληροφορίες για τους χρήστες των εξοπλισμών αυτών, σημεία αναφοράς και εκστρατείες ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση, ε, την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών. Έχω μια ε, μόνη αντίρρηση, μόνο μια επιφύλαξη γιατί αναμένω feedback, ε, ενημέρωση δηλαδή από πλευράς του κλάδου ώστε να κατανοήσω καλύτερα πώς και αν αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν πράγματι να ε, λειτουργήσουν από δικητική διοικητική άποψη. να ευχαριστήσω λοιπόν ακόμα μια φορά την εισηγήτρια για την ε, ε, εξαιρετική της εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλας από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα που είναι αρκετά τεχνικό. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους. Ανησυχούμε ότι αν κάτι είναι ε, ελαττωματικό, ε, οι ανθρώπινες ζωές διακυβεύονται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς ε, θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το ζήτημα. Κάτι που πρέπει να επισημάνουμε. Εμείς μόνο γνωμοδοτούμε για το θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι σωστό γιατί ε, είναι σημαντικό να ακουστεί περισσότερο η άποψη των εργαζομένων. Υπάρχει μια οδηγία σήμερα και υπάρχει μια πρόταση για κανονισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να οδηγούν στο γεγονός ότι απλοποιείται με την νομοθεσία αλλά επεκτείνεται και το πεδίο εφαρμογή της γιατί υπάρχουν και μερικά μεμονωμένα προϊόντα τα οποία θα ε, διέπονται πλέον από αυτόν τον ε, κανονισμό. Κάτι άλλο που μου φαίνεται επίσης ε, σημαντικό Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε γενικέ γραμμές βέβαια με τη βάση της συζητήτριας. Στην ΙΜΚΟ η πρόεδρο, ε, η Βίκη Φόρντ, διέγραψε ένα από τα στοιχεία που για μας είναι μία πρόοδο και μία ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ε, δηλαδή ότι όλα αυτά τα προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα, να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει καλύτερος έλεγχος της ποιότητας. Υπάρχει μία πρόταση από πλευράς Προέδρου Ίμκο για διαγραφή. Δηλαδή αυτή η έγκριση ε, θα είναι εσαΐ ε, ε, χωρίς έλεγχο. Εμείς νομίζουμε όμως ότι ε, νομίζω ότι αυτό είναι λιγότερο καλό από την πενταετή αναθεώρηση. Υπάρχει Υπάρχει βέβαια η ιδέα του ελέγχου, αλλά δεν υπάρχει ο πενταετής έλεγχος. Εμείς προτείνουμε να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Δεύτερον, είμαστε αρκετά ανοιχτοί στο γεγονός ότι κάποιοι τομείς ε, βιομηχανικοί ε, να ελέγχονται κάθε χρόνο και το γεγονός ότι θα πρέπει εκτός από αυτόν τον ετήσιο έλεγχο και κάθε πέντε χρόνια καινούριο έλεγχος, αυτό θα ήταν, αυτό θα ήταν αντιθέτως υπερβολή. Εκτός λοιπόν από αυτά τα δύο σημεία που για μα είναι <clears throat> ε, σημαντικά, νομίζουμε ότι ε, και η δουλειά της ΙΜΚΟ και η δουλειά της ε, εισηγήτριας της δικής μας πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λαμπάγεβα. Ντλαμπάγεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέλους της συναδέλφου θα ήθελα να πάρω το ε, λόγο Τρεις στόχους ε, πιστεύω ότι έχει αυτό το κείμενο είναι να βελτιώσει τη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας όπως επίσης και να εξασφαλίσει ένα ισότιμο πεδίο ε, για τα μέσα αυτά. Οι οικονομικοί φορείς ε, των οικονομικών φορέων εντός της εσωτερικής αγοράς όπως επίσης και καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον στον τομέα των ατομικών μέσων προστασίας. Κατά την άποψή μα, η Επιτροπή μας θα έπρεπε να επικεντρωθεί κυρίως στην πτυχή της ε, εργασίας ε, με ε, ενίσχυση της ασφάλειας και της υγεία των πολιτών. Δεν θα έπρεπε να, να επικεντρωθούμε περισσότερο στις λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι δουλειά της ΙΜΚΟ Είμαστε λοιπόν μιας ε, πιο στοχοθετημένης προσέγγισης και για τους χρήστες ε, ατομικών μέσων προστασίας ε, να υπάρχει καλύτερη εξασφάλιση. Εγώ χαίρομαι, Λάουρα, που έχεις δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τελικό χρήστη των μέσων αυτών, γιατί πιστεύω ότι ο, ο, άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και πρέπει να είναι το σημείο εστίασης της εργασίας μας. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως σε μια στοχοθετημένη προσέγγιση, γιατί η περίπλοκη νομοθεσία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητες συνέπειες και μπορεί τελικά να μην ε, επιτύχουμε το στόχο προστασίας των εργαζομένων. Κάτι ακόμη σημαντικό και πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό είναι η απλοποίηση της νομοθεσίας και η εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι δυσανάλογος ο βαθμός που πλήττονται από την περίπλοκη νομοθεσία γιατί δεν έχουν τους σπόρους να την αντιμετωπίσουν, κάτι το οποίο έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτές θα είναι τουλάχιστον ε, τα δικά μας κριτήρια για τη δική μας δουλειά και ε, σε αυτά τα στοιχεία θα βασιστούμε κατά την υποβολή τροπολογίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της ως τώρα και ε, εναγωνίως περιμένουμε την ε, συνέχεια της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Μάκεντάιρ από την ECR. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την ησυχήτρια. Ε, Λάουρα, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ σκληρή δουλειά σου. Την εκτιμούμε ιδιαίτερος ε, και αναμένουμε εναγωνίως τη συνεργασία μαζί σου προς ένα καλό αποτέλεσμα η τρέχουσα νομοθεσία για τα ατομικά μέσα προστασίας χρειάζεται ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό είναι το πακέτο μέτρων που σκοπό έχει να ευθυγραμμίσει ε, και να απλοποιήσει την νομοθεσία σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Πρέπει βέβαια να έχουμε ε, ισχυρές απαιτήσει σε σχέση με τα ατομικά μέσα προστασίας, όμως αυτή η πρόταση ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον εξυγχρονισμό και την απλοποίηση μια, ενός ήδη ε, ε εύρυθμα λειτουργούν συστήματος και επομένως δεν νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολλέ αλλαγέ. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι είναι αποτελεσματική η νομοθεσία, όμω πρέπει να αποφύγουμε και την κατάσταση κατά την οποία με τι καλύτερε των προθέσεων θα καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα το οποίο θα είναι πολύ βαρύ, ε, δυσανάλογο και δεν θα εξυπηρετεί και το στόχο μας. Οπότε πρέπει να εξεύρουμε μια ισορροπία και πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις ε, να συμμορφώνονται με μια νομοθεσία που θα είναι σαφής, απλή και αποτελεσματική. Ο ρόλος μας ως συνομοθετών λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης και δεν εννοώ καμία νομοθεσία, εννοώ ότι πρέπει να έχουμε απλούς νόμους, απλούς κανόνες, ε, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις κυρίως να μπορούν να συμμορφωθούν γιατί καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν και νομίζω ότι η διαχείριση του κινδύνου και η τα επιστημονικά στοιχεία πρέπει να είναι η βάση για την ασφάλεια και την υγεία σε κάθε ε, ενωσιακό ε, κανονισμό. Εμείς θα υποβάλουμε κάποιες τεχνικές τροπολογίες, δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες εδώ. Υπάρχει κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε και είναι το εφικτό της ε, πενταετούς μέγιστης εγκυρότητας της πιστοποίησης. Έχουμε ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι είναι πολύ μικρή αυτή η χρονική περίοδος δεδομένου του κύκλου ζωής των συγκεκριμένων μέσων προστασίας. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό όταν θα κάνουμε λεπτομερέστερη συζήτηση στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Όσον αφορά τώρα τη χρήση του ίντερνετ, των iPhones και τη πλήρη χρήση της ε, ε, τεχνολογίας εχμής, νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, ώστε να ενημερώνεται καλύτερα το ε, εργατικό δυναμικό μας για, το, για τη χρήση αυτών των μέσων προστασίας. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ Λόρα για την δουλειά σου ως τώρα και αναμένω τις συζητήσεις στις συναντήσεις για τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τατσιώνα Στανόκα από τους Πράσινους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κύριου Ρέντκε, της κυρίας Ρέντκε που είναι ε, σκιώδης αλλά δεν μπορεί να παραστεί σήμερα στη συνάντησή μας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, στους συναδέλφους ορισμένα στοιχεία για τη σημασία αυτών των μέσων ατομικής προστασίας. Το 2007 υπολογίστηκε ότι 23 εκατομμύρια εργάτες είχαν ε, προβλήματα που σχετίζονταν, υγείας που σχετίζονταν με τον χώρο εργασίας. Το 2011 έγιναν 2,7 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα που κατέληξαν σε περισσότερες από τρεις μέρες απουσίας από το χώρο εργασίας και το και 30.000 306.000 ε, ε, θανατηφόρα ε, εργατικά ατυχήματα έγιναν στους χώρους Από αυτή την άποψη είναι σαφές πόσο σημαντική αρκεί για την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των ανθρώπων είναι αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας. Η χρήση τους είναι απαραίτητη για να μειωθούν τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας. Και πρέπει να εξασφαλιστούν μεχανισμοί ελέγχου και επιτήρησης ε, μετά τη διάθεση τέτοιων μέσων ατομικής προστασίας στην αγορά. Και όποτε υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει ο κατασκευαστής να ανακαλεί τα προϊόντα από την αγορά. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την κατάλληλη χρήση θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και οι οδηγίες θα πρέπει να είναι ευσύνοπτες και όσο το δυνατόν σαφέστερες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αδήλωτη εργασία. Γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα αυτό όσον αφορά την ασφάλεια ε, ε, στην εργασία και έτσι ε, οι εργάτες εκτίθενται σε υψηλούς κινδύνους και δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Επίσης, οικιακές δουλειές που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες δημιουργούν και σχετίζονται με ιδιαίτερους κινδύνους και Υποστηρίζοντας λοιπόν το έργο της εισηγήτριας ως ομάδα και τις ε, τροποποιήσεις που θα υποβάλει στο σχέδιο κανονισμού θα ε, υποβάλουμε και εμείς ορισμένες τροποποιήσεις για αυτή την αδήλωτη εργασία και την ενδεδειγμένη χρήση, συντήρηση και τον καθαρισμό των μέσων ατομικής προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η Ίνες Τσούμπερ από την ομάδα Γκούε. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί έτσι μπορούμε να προετοιμαστούμε για τις ψηφοφορίες και να τις ξεκινήσουμε. Απλά να αναφέρω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών για αυτήν την έκθεση για τα μέσα ατομικής προστασίας είναι η 3η Μαρτίου 12 η ώρα το μεσημέρι και η έγκριση στην ε, ε, Επιτροπή μας θα γίνει την 1η Απριλίου 2015. Πάμε στις ψηφοφορίες. then we'll start the voting. Ωραία, ξεκινάμε με τις προφορίες. Πρώτα έχουμε το Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και για ε, την υποστήριξη προς τις δραστηριότητες της ε, εταιρείας ε, Attica Publishing στην Ελλάδα. Το ΕΛΚ έχει έναν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Εξακολουθεί το ΕΛΚ να έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ακόμη. Παραμένει το πρόβλημα. Ξεκινάμε από την αρχή. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Πάλι. Ένας παραπάνω. Συγγνώμη. <laughs> yes. <laughs> Did you find him or her? <laughs> still sorry to say, but we go Παραμένει το πρόβλημα, είναι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Now it's, okay. The vote is... Ωραία. Τώρα εντάξει, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Και περνάμε στο θέμα της Attica Broadcasting στην Ελλάδα, ένας ψηφοφορία. Are there Πέρας. Εγκρίνεται. Κύριε Κάσα. Ε, κύριε Πρόεδρε, πρωτού περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Το ΕΛΚ συμφωνεί με το κείμενο της προφορικής ερώτησης όπως έχει διατυπωθεί. Αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι ε, ο καλύτερος χρόνος, μιας και η Κομισιόν περιμένει ακόμα ορισμένε προφορίες από τις γερμανικές αρχές. Και στο πλαίσιο αυτό ε, προτείνουμε την αναβολή την, ε, της προφορίας για την έγκριση της συγκεκριμένη ε, προφορικής τροπολογίας. Ε, ε, ε, Μα δεν αποτελεί ε, αμυγός γερμανικό θέμα η ε, καθιέρωση των ορίων αποδοχών. Μιλάμε για μια τοποθέτηση επί της αρχής. Γι' αυτό ε, εμάς, άποψή μας είναι να παραμείνει το θέμα στην ημερήσια και να γίνει σήμερα η ψηφοφορία. Κυρία Χάρκιν, πολύ σύντομα να πω ότι συμφωνούμε με το ΕΛΚ. Θεωρούμε και εμείς δηλαδή ότι αν, αν, υπήρξε, αν υπήρχε απάντηση από την Κομισιόν και νομίζω ότι οι γερμανικές αρχές θα δώσουν τις πληροφορίες 4 Μαρτίου. Αν θα είχαμε τότε μια απάντηση ε, και θα ήταν καλύτερα να θέσουμε τότε την, ε, την ερώτησή μας. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να το κάνουμε τότε. Ε, από την άποψη δηλαδή του timing, ίσως όντως θα συμφωνήσουμε και εμείς με το ότι θα ήταν καλύτερη η αναβολή μιας τέτοιας για την ΚΟΕ. Καλημέρα σας. Εμείς θα θέλαμε τώρα να ψηφιστεί αυτή η προφορική ερώτηση. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή το θέμα για τον τομέα τούτο και όπως ήδη υπόθηκε επηρεάζει ολόκληρο τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. E η κυρία Μάκιντάιρ από το ECR. Συμφωνώ με το, με το ΕΛΚ και με την ε, Χάρκινγκ. Δεν θα, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε, συμφωνώ απολύτως. Οπότε, λέει η Πρόεδρος, για να, να ψηφίσουμε, για να είμαστε τυπικοί ηλεκτρονικά, για το αν θα γίνει σήμερα ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, ποιοι είναι υπέρ της αναβολής της ε, ψηφοφορίας. Ένας ψηφοφορίας. Ψηφίσαν όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Okay, then we'll vote. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα τελικά. Έχω το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας. Ψηφοφορία επί της ερώτησης προς την Κομισιόν ξεκινά λοιπόν η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Now we'll vote on uh, the draft report by Mr. Να ψηφίσουμε τώρα για το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Γκουτιέρε Πριέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Ξεκινάμε με την τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχή, αποχές εγκρίνεται. Μάλλον ας ψηφίσουμε ε, ηλεκτρονικά. Ένας ψηφοφορής. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση L υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ένας εξωφορίας συμβαστική πρόταση L έναρξη εξωφορίας τέλος της προφορία εγκρίνεται Then we end up at compromise M. Συμβαστική πρόταση M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 109, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ολοκληρωτικά για την τροπολογία 110. The vote is open and now the vote is closed. Ένας και τέλος της φοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας Εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Καταπίπτει. Α, ναι. Πάμε στην τροπολογία 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 120 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 121. Θα ψηφίσουμε αργότερα για την τροπολογία αυτή και θα περάσουμε στην τροπολογία 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση έν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένας ψηφοφορίας πέρας ναι, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση O. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 140. Είναι η επόμενη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορίε. Πέρα ψηφοφορίε. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική πρόταση π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 152 κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 150, τροπολογία 150, ένας ψηφοφορίας, λήξη ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 151, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 154 θα την ψηφίσουμε αργότερα. Περνάμε στην συμβαστική πρόταση Q, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 157. τη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 158. Να πω μόνο ότι αν εγκριθεί σημαίνει ότι καταπίπτει η συμβαστική πρόταση R. Ψηφίζουμε για την 158 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στη συμβαστική πρόταση R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση S υπέρ κατά την εγκρίνεται. Τροπολογία 175 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Αποχές και εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση U, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 189 ε, υπέρ, κατά, Εποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να το ελέγξουμε. Ένα ψηφοφορία. Λήξη. Τη υποφορία για την τροπολογία 189. Συμβαστική πρόταση Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση W υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην ψηφοφορία για την τροπολογία 200, υπέρ, κατά, αποχές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορίας. Και τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 201 καταπίπτει. Περνάμε στη 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 203 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για 205 ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. Ναι, απορρίπτεται όντως. Τροπολογία 206 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική πρόταση έξ, υπέρ κατά αποχές Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Άγγια. Ε, σε Αν μπορεί κάποιος να επαληθεύσει εδώ τη λειτουργία των ε, μηχανημάτων για την ψηφοφορία. Α, έχετε πρόβλημα με το, με το μηχάνημα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει. Check that you have your card uh, down all the way. We are on. six. We go back to compromise X. Ε, those in... Πάμε στην ε, πρόταση έξ, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 219. Ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα και τέλειωσε η ψηφοφορία. Yeah, Εγκρίνεται. Μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 220 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση Why. Uh, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 235, στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 236, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση Z. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 244, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ε, μπορώ να κρίνω με το μάτι, γιατί σηκώσατε πολύ λίγο το χέρι σας. Ξεκινάει η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...253, τροπολογία 253 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 254 και 255 και 56 θα ψηφιστούν μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις τρεις τροπολογίες, 254, 55 και 56. Ξεκινάει η ψηφοφορία και λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 2.58 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 2.58. Παρακαλώ, ναι. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 2.58. Σοφία Ριμπέιρο, Χάιντς Μπέκερ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 259. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 264. Αν εγκριθεί η συμβαστική πρόταση ΑΑ θα καταπέσει. Αλλά πρώτα θα ψηφίσουμε ε, για την τροπολογία 264. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Οπότε περνάω στη συμφορία για την συμβαστική πρόταση ΑΑ, AA, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση ΑΒ, AB, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 289, τροπολογία 289, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την 289 ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 290 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία όχι, θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 290. Ένα ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 33 ψήφου υπέρ. Τροπολογία 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορία. Πέρσοφορες της ψηφοφορίας. Ο, απορρίπτεται. 2.92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση AC. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε για την 302 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 303, για την τροπολογία 303. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Ναι, απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μάλλον θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένας ψηφοφορίας. Και τέλος της ψηφοφορίας. Για την 304 πάντα, ναι, ναι. Εγκρίνεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημά σας. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 304, για την τροπολογία 304. Εντάξει, θα το ξανακάνουμε λοιπόν. Ξεκινά τώρα η ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε, για την τροπολογία 304, 304, Πέρασε της ψηφοφορίας, τώρα δεν υπήρξε πρόβλημα, ωραία, εγκρίνεται. Τροπολογία 305, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 306, υπέρ, Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 305. Ωραία. Ένας ψηφοφορίας για την τροπολογία 305 και πέρα ψηφοφορίας. Yes, it's carried. We go... Εγκρίνεται. Λοιπόν, 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AD υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 317 υπέρ. Κατά νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε καλύτερα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. 318. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε τώρα στην 321 για διαγραφή Φυσικά αν ισχύει αυτό καταπίπτει ο συμβιβασμός. Ψηφίζουμε λοιπόν την 321 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΕ e, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AR στο Τέλος της σελίδας υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε

γιατί εγκρίναμε τη συμβιβαστική AE. Πάμε λοιπόν σε 325 τώρα, υπέρ. Α, το ίδιο ισχύει και για την 325. «327 είναι η επόμενη που θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 336 υπέρ κατά αποχές. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε γιατί δεν έβλεπα καλά τα χέρια σας. Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 336. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε. Στην 343. Έχετε το λόγο κύριε Κουτιέρη. Πρέπει να ψηφίσουμε την 327. Τη Βερόνικα Λόπ Φοντανιέ. Μα την ψηφίσαμε και, και εγκρίθηκε. Now 343 343. Κάτω-κάτω στη σελίδα 26. Υπέρ. σελίδα 26, τροπολογία 343. Συγγνώμη, εσείς έχετε άλλη, άλλο έγγραφο ίσως. Λοιπόν, τροπολογία 343, Μαρία Ρένα και Μπαγιέ Λοιπόν, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Άρα ψηφίζουμε την 346 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 346, ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας. Εγκρίνεται. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 356 της Μόνικα Βάνα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε, εντάξει, 357, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 358. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 359. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίπτεται 360 υπέρ κατά Α, αποχές. Εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 362. Αποσύρεται. 365. Οι 363 και 365 είναι ταυτόσιμες. Ήθελα να πω απλώς ότι αν ψηφιστούν, καταπίπτει ο συμβιβασμός. Ψηφίζουμε λοιπόν την 363 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 365 είναι ταυτόσημη. Οπότε πάμε στη συμβιβαστική AH. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 371 έχει καταπέσει. 373 άρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AI. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AS. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα πάμε στην 387. Στην επόμενη σελίδα υποθέτω για τους περισσότερους υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 388 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 390 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93, 91 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Καλώς. 391. Έναρξη. Πέρασα. Εγκρίνεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα έξι τροπολογίες από την 392 ως και την 397. Όλες αυτές είναι ταυτόσιμες. Αν υπερψηφιστούν, τότε η συμβιβαστική AJ καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα αυτές τις τροπολογίες όλες μαζί, 392 με 397 όλες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άρα συμβιβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος της 405. Υπέρ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 407. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 409. Αν θέλετε να ελέγξουμε τη 407. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορία για τη 407. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 409. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 408. Κάποιος ήθελε να ελέγξουμε την 409. Ελέγχουμε την 409. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 408 καταπίπτει, άρα 410. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ε, ε, ε, Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική AL υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε την 423. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 424. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 425. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 426 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 427 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AM. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 442. Υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 443. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική AO. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα πηγαίνουμε Μισό λεπτό. Καταπίπτει. Άρα πάμε στην 448. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 452 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 453 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο Τη 453. Ωραία, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίψετε. Συμβαστική AP. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 462. 462 λοιπόν, υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 463 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 464. Αν υπερψηφιστεί, τότε η συμβιβαστική παρακάτω, AQ, καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AQ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 472 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 472. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Α, ένα μηχάνημα του ΕΛΚ δεν δουλεύει. Έχει προβλήματα, έχετε προβλήματα με το μηχάνημα. Κοιτάξτε, δεν θα τσακωθούμε. Να ξανακάνουμε τη ψηφοφορία, τι να πω. Έναρξη. 472 ψηφίζουμε. You understand that you... Yes, you have to push the button, yes. Πρέπει να το πατάτε το κουμπάκι. Λοιπόν, ψηφίσαμε. Λοιπόν, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Μέχρι και την 7. Τη ψηφίζουμε όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Πάμε τότε στη συμβαστική A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά. Covered by the compromise, so it's not, it's not Okay. It's not Then we vote... Ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 13 που δεν καλύπτεται το συμβιβασμό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Έλεγχος της 13. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Να ξαναρχίσουμε. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Και πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ή. E. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 48. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 49. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται, να. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος της 50. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, συγγνώμη δεν μου είναι σαφές έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λοιπόν την 72. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικής. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΆΙ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 τώρα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Να ελέγξουμε την 85. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Ηλεκτρονικός, ηλεκτρονικός θα το ψηφίσουμε. Άρα έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 38 υπέρ, 10 κατά. Τελείωσε ο κατάλογος της ψηφοφορίας μας και η ηλεκτρονική, η ηλεκτρονική μας ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Sorry, there was some sort of mistake. Συγγνώμη, έγινε κάποιο λάθος με τους αριθμούς. Με την τελευταία ονομαστική ισοφορία. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Πρέπει να γίνει ψηφοφορία για άλλη μια τροπολογία. Ε, συγκεκριμένα πρέπει να επαναλάβουμε την τελευταία ψηφοφορία που κάναμε. our new uh, Είναι νέα απόφαση για τη διαφάνεια ώστε να ξέρουν οι ψηφοφόροι μας πώς ψηφίζουμε, πώς ψηφίζει ο κάθε ευρωβουλευτής εδώ στην αίθουσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ε, ε, επαναλάβουμε την ε, τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Πρέπει να έχετε τις κάρτες σας λοιπόν. ονομαστική ψηφοφορία για, για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ένας ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλεια. Θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν. Είναι σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. 38-10. Και τώρα πλέον ξέρουμε πώς ψήφισε ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ Okay, friends. Uh, we'll start. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. the meeting. Ε, Ωραία, προχωράμε με το επόμενο θέμα μας και δίνω το λόγο για να μας μιλήσει για μια πολύ σημαντική έκθεση ο κύριος Μπέκερ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόληση, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίε κινητικότητα και περαιτέρω ενοποίηση των Εργαζομένων εργασία. Ο λόγο στον κύριο Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία της Κομισιόν. και οδήγησε σε πολύ ενεργή συμμετοχή των ευρωβουλευτών, 699 τροπολογίες. Κατά τη γνώμη μου, τα παρακάτω είναι τα βασικότερα ζητήματα που τίθεται. Πρώτον, η συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων ως προς το αντικείμενο της ε, έκθεσης και η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, η συνεργασία με τα εθνικά γραφεία συντονισμού και τους κοινωνικούς εταίρους η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στην ομάδα συντονισμού και, και κατά τον ε, σχεδιασμό του προγράμματος. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους είναι απαραίτητη η εμπειρογνωμοσύνη και η διαβούλευση, οι γνώσεις των κοινωνικών εταίρων είναι απολύτως κάθοριστική σημασίας και θεωρώ ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη ε, δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά η συμμετοχή τους ε, στη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικά, σημαντική. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα, οι διασυνορικές εταιρικές σχέσεις, δηλαδή η δραστηριοποίηση του δικτύου Γιούρες στα διασυνοριακά θέματα. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι είναι και θα προσπαθήσω να το εντάξω στην έκθεσή μου. Στο, υπάρχει ένας τρίτος τομέας όπου υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και μιλώ συγκεκριμένα για την ε, ενσωμάτωση θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο δίκτυο Γιούρες. Ε, Θα πρέπει και να απαιτήσουμε την ένταξη τέτοιων ε, θέσεων πρακτικής άσκησης, αλλά και να τεθούν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό αυτή η πρόθεση είναι θετική, συμφωνούν και πολλοί συνάδελφοι μαζί μου, αλλά αφού ξεκινούμε τις ε, διαπραγματεύσεις μας και τις, ε, την προσπάθεια εξέβεσης συμβιβασμών, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά θέματα όσον αφορά το αν θα είναι προϋπόθεση να ε, να είναι η σύναψη κανονικής ε, σύμβασης εργασίας. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για προσθήκη ή και αφαίρεση εταίρων από το γιούρος. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα και να προστίθενται εταίροι στο γιούρος αλλά και να απομακρύνονται από το γιούρος. Έχουμε και μια πρώτη εικόνα ε, για τις ε, εκτελεστικές και τις ε, κατεταξιδότητες πράξεις. Θέλουμε η Κομισιόν να μην μπορεί να αποφασίζει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά από την άλλη πλευρά πρόκειται και για ένα ζήτημα το οποίο συμπεριλαμβάνει και μια σειρά τεχνικές διαστάσεις χωρίς πολιτική σημασία. Θα το εξετάσουμε βεβαίως και αυτό το θέμα και σε συνεργασία θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Επίσης, θέλω τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων και να μην ακούγεται απλώς η γνώμη τους. Θεωρώ ότι η δημοσίευση θέσεων απασχόλησης από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, είναι μία από τις δυνατότητες, αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσον αφορά την σύνταξη ε, αξιολόγησης ετησίως, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι ε, θετικό. Θα πρέπει όμως σε πρώτη φάση να προβλεφθεί να, μια ε, φάση πρώτης εφαρμογής. Υπάρχει και το ζήτημα της ε, μετέπειτα αξιολόγησης, της αξιολόγησης σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν, τα σχόλια που έχω λάβει είναι πολύ θετικά Επίσης υπήρξε πρόταση να αντικατασταθεί ο όρος εργατικό δυναμικό με, τους, με τον όρο αναζητούντες, άτομα αναζητούντα εργασία. Θεωρώ ότι είναι θετική και αυτή η πρόταση. Επίσης υπήρξαν και κάποιες παρατηρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ε, γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των ε, κρατών μελών. Αν δείτε τα άρθρα 45 και 47 υπάρχουν διάφορες διατάξεις για θέματα που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε εδώ. Και μιας και βρισκόμαστε στην έναρξη των ε, συζητήσεων θα ήθελα να σας πω από τώρα ότι είμαι ανοιχτό στο να εντάξω και να αποδεχθώ τροπολογίες εφόσον όμως ενισχύουν οι τροπολογίες αυτές την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας εφόσον δεν ενισχύουν το γραφειοκρατικό φόρτο και δεν αποδυναμώνουν το δίκτυο Γιούρες. Σκοπός μου είναι σε συνεργασία με τους σκιώδεις να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας από τις 10 Μαρτίου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα γιατί πρέπει να κάνω, ε, έχω ένα ταξίδι που πρέπει να κάνω την επόμενη εβδομάδα ε, ως ε, εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Σε κάθε περίπτωση θα σας δώσω το πρόγραμμα εργασιών που θέλω να ακολουθήσουμε. Να σας ευχαριστήσω βεβαίως για άλλη μια φορά για τις ε, εξαιρετικά πολύτιμες τροπολογίες που ε, υπέβαλαν ε, όλοι οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Μπέκικερ. Ο λόγος τώρα στους σκιώδεις συζητητές. Να πω και εγώ κάποια λόγια. Ένα μέλος της γραμματείας, η Κάλια Σέβεριν. Σηκωθείτε παρακαλώ για να σας δούμε. έχει επιδείξει ε, μεγάλο επαγγελματισμό και δυστυχώς ε, θα μας αφήσει, θα φύγει, θα πάει να δουλέψει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, Οικονομικών Υποθέσεων. Οπότε νομίζω ότι της αξίζει ένα χειροκρότημα για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Ευχαριστώ Κάγια και ελπίζουμε τα ζητήματα απασχόλησης να λαμβάνονται πιο πολύ υπόψη στις εργασίες της Επιτροπής ε, ε, Οικονομικών Υποθέσεων. Ο Σον Σάιαν έχει το λόγο εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Σας συγχαίρω για το γεγονός ότι ηγηθήκατε αυτής της διαδικασίας. Και από την πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε ότι θα έχετε τη συνεργασία μας. Προς το παρόν μπορούμε θεωρώ να κάνουμε βήματα στη σωστή κατάσταση ακόμη και αν δεν καταργήσουμε βεβαίως την εκμετάλλευση και όλα τα προβλήματα. Αυτό που με εξέπληξε μελετώντας τη συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν είναι το πώς η, η μεγάλη απουσία ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως, του, ως προς τους ε, ορισμούς. Δεν υπάρχει κοινός ορισμός για το τι είναι η εργασία, τι είναι η μαθητεία, τι είναι η πρακτική άσκηση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία θέλουμε να, να ε, εμβαθύνουμε. Πώς μπορούμε αλλιώ να θεσπίζουμε νομοθεσία αν δεν έχουμε κοινού ορισμού. Θα επισέλθω αργότερα σε πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Επίσης, το όλο πλαίσιο βασίζεται στην ε, αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στα κράτη-μέλη. Αλλά η αποτελεσματικότητα αυτή δεν σημαίνει ε, λογοδοσία των υπηρεσιών αυτών. Οπότε, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στους τομείς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προσωπικά ε, υπέβαλα 54 από τις 699 τροπολογίες. Δεν θα μιλήσω για τις δικές μου τροπολογίες. Ε, ξέρω ότι όλοι σας ξενυχτήσατε χθε ε, το βράδυ για να τις διαβάσετε και έχετε εικόνα, αλλά ε, θα αξιοποιήσω το χρόνο που μου δίνετε για να θέσω κάποια ερωτήματα για τροπολογίες που έχουν επιβάλει άλλα μέλη της Επιτροπής που πράγματι ξενύχτησα για να τις ε, διαβάσω και για τις οποίες έχουμε σχηματίσει έχουμε εικόνα για τις πρακτικές ασκήσεις ε, και, την, και την μαθητεία για την τροπολογία 306 από το ΕΛΚ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπέκερ και τους συναδέλφους του ΕΛΚ πώς θεωρούν ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητευόμενοι στους οποίους θα προσφέρεται εργασία θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα ως εργαζόμενοι. Και για την 292 ε, τροπολογία από, την, από τους φιλελευθέρους να μας πούν τι εννοούν όταν λένε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να διέπει τις πρακτικές ασκήσεις και τις μαθητείες. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος ευρωπαϊκός. Δεν αναφέρονται πουθενά αυτά τα δύο θέματα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν θέλουμε φυσικά να αγνοήσουμε τα ζητήματα αυτά, αλλά δεν θέλουμε επίσης οι νέοι άνθρωποι να γίνονται ε, αντικείμενο εκμετάλλευσης. Επίσης, δεν έχω κατανοήσει ακόμη αυτή τη διάκριση που κάνουν άλλες ομάδες για τους εταίρους και τα μέλη του Γιούρες. Στην 208 ε, του ECR οι εταίροι ε, ταυτίζονται με τις υπηρεσίες απασχόλησης, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ε, πολύ λογικό. Δεν είναι ε, πολιτικού χαρακτήρα αυτή η διάκριση. Από τεχνικής άποψης, αν θέλουμε να θεσπίσουμε ε, ένα νομοθέτημα, θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Για την τροπολογία που υπέβαλε η ε, Γκουεν για τα τέλη, Έχουμε συμφωνήσει όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν θέλουμε να υπάρχει χρέωση. Μπορεί μήπως η Γκουέ να μας εξηγήσει γιατί εκείνη επιλέγει κάτι τέτοιο. Και για το άρθρο 14 που νομίζω ότι είναι το κεντρικό άρθρο του όλου εγγράφου όπου ορίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να ε, ανακοινώνουν όλες τις κενές θέσεις εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης τους στο Γιούρες. Έχουμε συμφωνήσει σε γενικές γραμμές με τον κύριο Μπέκερ και για να το ξεκαθαρίσουμε, το σύστημα όπως έχει σήμερα δεν λειτουργεί. Υπάρχουν ε, ένα εκατομμύριο και θέσεις εργασίες από, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 650.000 από τη Γερμανία, 300.000 από την ε, Ιταλία. Δεν πρόκειται, δηλαδή με άλλα λόγια, για ένα αποτελεσματικό σύστημα που να ενισχύει τις αδελφικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιτνάνσκα από το ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπέκερ. Νομίζω ότι η συνεργασία μας μέχρι στιγμής ήταν υποδειγματική. και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Προσωπικά έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα ενεργά και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη αυτού του συστήματος. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπέκερ στην τελευταία μας ε, συνάντηση. Είναι σημαντικό να γίνει γνωστότερο στην ε, κοινή γνώμη το συγκεκριμένο ε, σύστημα, το συγκεκριμένο δίκτυο. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανεργία και γενικά, αλλά και ε, όσον αφορά συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αμαία, περιοθεροποιημένες κοινωνικές ομάδες. Είναι σημαντικό και τα μέλη αυτών των κοινωνικών ομάδων να μπορούν να αξιοποιήσουν την κινητικότητα των εργαζομένων και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ε, καταργηθούν τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι στιγμής στο ε, Θα πρέπει και τα άτομα με αναπηρίες, λοιπόν, να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο δίκτυο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έχω συγκεκριμένες, συγκεκριμένη εμπειρία από την ε, ε, Σλοβακία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Θα πρέπει εκ των προτέρων όλοι να γνωρίζουν τι και πώς λειτουργεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι τα, οι εταίροι και τα μέλη θα πρέπει να έχουν διαφορετική θέση εντός του δικτύου, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν για το ε, ποιος θα αποτελεί μέλος, ποιος θα αποτελεί εταίρο και ταυτόχρονα θα πρέπει στον κανονισμό να ενταχθούν τα εξής στοιχεία. Όταν και εφόσον κάποια ιδιωτικά γραφεία έβρεσης εργασίας πληρούν κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις, θα πρέπει να υπάρχει νομική ε, ασφάλεια. Αν κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορεί να γίνει μέλος. Αν δεν πληρεί τις ε, προϋποθέσεις, τότε δεν θα πρέπει να μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει δηλαδή, όπως είπε και ο κύριος Μπέκερ, ε, να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης μελών ε, στο Eures, αλλά και αφαίρεσης μελών από το Eures. Και χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που θα συνεχιστεί σίγουρα και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους υπόλοιπους ε, σκιώδες για τις παρατηρήσεις τους και για πολύ καλή συζήτηση. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ένωση είναι σημαντικός παράγοντας για να αντιμετωπιστεί η ανεργία κυρίως αυτή των νέων. Γι' αυτό και θα πρέπει ταχαία, ταχαίως να υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός. Ε, πιστεύω θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και να κινηθούμε γρήγορα. Όλοι συμφωνούμε ως κοιόδης εισηγητές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σύγχρονο δίκτυο ε, θα είναι ε, γνωστό και αποτελεσματικό στους πολίτες, για τους πολίτες της Ευρώπης. Εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχήν θα πρέπει να δίνονται, να δίνονται οι διαθέσιμες θέσεις ε, αλλά και οι δυνατότητες για μαθητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ε, περιορίσουμε τις, τις ε, θέσεις εργασίας στα είδη συμβάσεως. Θα πρέπει να μπορούν οποιαδήποτε είδος απασχόλησης να βρίσκουν. Είτε είναι μαθητεία είτε είναι κανονική σύμβαση. Να ενθαρρύνουμε τους αναζητώντες εργασία και κυρίως τους νέους γιατί ότι αυτοί είναι πιο ε, ε, πιθανό να κινηθούν για να εργαστούν. Οι θέσει θα πρέπει να είναι επίση ανοιχτέ για όλου όσου έχουν το νομικό δικαίωμα να εργάζονται στην Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιο είδους ε, θέσεις ε, όπου θα χρειάζεται μια κεντρική ας πούμε, ηθαγένεια για, ας πούμε, για θέσεις που έχουν να κάνουν με την κρατική ασφάλεια. Διαφορετικά πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους όσους έχουν δικαίωμα να εργάζονται στην Ένωση. Εγώ θα άλλαζα λοιπόν τη διατύπωση σε job seekers Έπειτα, το γιούρι θα πρέπει να είναι δωρεάν. Να είναι φιλικό προς το χρήστη, να μπορούν να παρέχουν δε υπηρεσίες και online και να είναι ε, προσβάσιμο για όλους. θα πρέπει να, υπάρχουμε, να, στοχεύσουμε σε διασυνοριακές εταιρικέ σχέσεις, ιδιαίτερα σε μέρη όπως ε, το δικό μου είναι πολύ σημαντικό και βλέπω και τους συναδέλφους από την Αυστρία και τη Σλοβακία. Πέμπτο η παρατήρηση. Ε, το να μπορέσει κανείς να παρέχει υπηρεσίες ε, είναι πολύ σημαντικό. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο ε, θα πρέπει ωστόσο να είναι και ελκυστικό να μπουν σε αυτό το σύστημα και να μην τους επιβαρύνει. Ε, θα πρέπει λοιπόν γρήγορα να κινηθούμε με την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού από το Ευρωκοινοβούλιο γιατί νομίζω πως η κατάσταση της αγοράς της Ευρώπης απαιτεί μεταρρυθμίσεις ε, για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη ελπίδα και ευκαιρίες απασχόλησης στους ανεργούς νέους της Ευρώπης. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις ηγητές για να την ολοκληρώσουμε την έκθεση και σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία μας τώρα. Σας ευχαριστώ η Παλώμα Λόπες. Ε, καλημέρα σας και ευχαριστώ. Ε, Καταρχήν να ευχαριστήσω για την εργασία την, ε, τον εισηγητή ε, και όλους όσους συμμετείχαν στη σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης. Έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες από πλευρά της ΓΟΕ που αφορούν πολλές και διάφορες πτυχές. Καταρχήν κινητικότητα. κινητικότητα δεν περιέχει θελοντικό στοιχείο, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου που επλήγησαν πολύ σοβαρά από την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν ακριβώς για να αντιμετωπιστεί η κρίση και που όπως είδαμε δεν λειτουργήσαν. Όπως λένε οι χώρες του Νότου, η κινητικότητα δεν είναι θέμα ε, εθελούσιο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο αυτή η κινητικότητα είναι θετικό στοιχείο από τη στιγμή που είναι καταναγκαστική λόγω της απώλειας ε, της θέσης απασχόλησης ή της αδυναμίας εξέβρεση νέα θέση απασχόληση. Έπειτα, δημόσιο τομέα δεν θα έπρεπε να καλυφθεί από ιδιωτικέ πρωτοβουλίε που εν γέννη από τι εμπειρίε που έχουμε για παράδειγμα στην Ισπανία ε, ε, παράγονται έτσι, δημιουργούνται μάλλον ε, ανισότητες που ιδιαίτερα για δύναμος ας πούμε ε, συμμετέχοντες ε, που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση. Το ίδιο και για τα πόρταλ που καθορίζουν τα αιτήματα ε, απασχόλησης ή τις θέσεις που προσφέρονται στο ίντερνετ. Δεν συμφωνούμε ούτε με την φόρους για τους εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα site το οποίο θα πρέπει να είναι δωρεάν έλεγχος και εποπτεία ε, για τους εταίρους αλλά και για το πακέτο μέτρων το οποίο θα πρέπει να ε, τεθεί σε εφαρμογή. Και τέλος, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο δραστήρια και ενεργή η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτήν τη, το δίκτυο ΕΟΡΕΣ για να μπορέσει να λειτουργήσει ορθά και για να μπορέσουν να αποφευθούν οι διακρίσεις όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank you, Jean Lambert from the... Ευχαριστώ, η Jean Lambert από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Εγώ μιλώ εξ ονόματος ε, του Τόμας Μάσερεκ που είναι ο σκιώδης για μας για αυτό το θέμα αλλά δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα. Να σχολιάσω ωστόσο κάτι προσωπικό διότι Απαντώ έτσι και σε κάποια από αυτά που υπόθηκαν. Ξέρουμε ότι ο κόσμος κινείται για λόγους ε, ε, εργασίας ε, αλλά και για διάφορους, με διάφορα αίτια. Ε, εμείς αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι στο Γιούρι η ποιότητα αυτής της εμπειρίας θα είναι όσο γίνεται πιο θετική σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Και αυτό είναι... αφορά και την πλευρά αναζήτησης της εργασίας όσο και την ίδια την εργασιακή εμπειρία. Και τώρα θα σας πω αυτά που θα λέγει ο Τόμας που λείπει σήμερα. Εμείς θα θέλαμε να είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό website αυτή η υπόθεση και ότι θα συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες και ότι το αυτόματο σύστημα αντιστοίχηση θα είναι αποτελεσματικό χάρη στις καινοτομίε. Πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του Γιούρες είναι η στήριξη της υπηρεσίας που δίνουν οι σύμβουλοι του Γιούρες και άρα τα μέλη να μπορούν να κατευθυνθούν σε πιο επαγγελματική ε, υπηρεσία ορατότητα και στήριξη στους συμβούλους του Γιούρις ώστε να παίξουν ρόλο κλειδί στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ε, λαμβάνουν αποφάσεις όντας ενήμεροι ε, για τα δικαιώματά τους για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, να έχουμε επίσης δυνατότητα ελέγχου με διάφορα μέσα, ας πούμε ε, συστάσεις αναχώρα που αναπτύσσονται από ε, τον Ευρωπαϊκό Εγωρισμό, να υπάρξουν περισσότερες συνεργασίες με εθνικά όργανα ελέγχου και ποιότητας. Δεν έχουμε δημιουργήσει νέα σώματα, αλλά ε, να υπάρξει πιο στενή συνεργασία και πιο καρποφόρα συνεργασία από αυτά, τα, ανάμεσα στους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν μέσω της οδηγίες για την απασχόληση, μετά στήριξη για την μάθηση ε, περισσότερων γλωσσών και ε, μη διακρίσεις ως ακρογωνίος λήθος για μια ομαλώς λειτουργούσα εργασιακή αγορά. Ε, ξέρω πως ε, οι σκιώδεις μας θα είναι πολύ ευτυχείς ε, ε, από τη συνεργασία με τον κύριο Μπέκερ και τους υπολείπους για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους χρήστες των, της υπηρεσίας Γιούρες. Ευχαριστώ. Λάουρα Αγγέα, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και κυρίως ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπέκερ. Ε, εύχομαι ότι οι που πρότεινα να μην ε, θεωρήθηκαν από το συνάδελφο ως ε, απλά και μόνο επικρίσεις. Εγώ θεωρώ πως εκεί που η Ευρώπη δίνει, παρέχει στοιχεία τα οποία αν χρησιμοποιηθούν καλά και με αποτελεσματικό τρόπο είναι θετικά θα πρέπει όντως να, να υπάρξει αυτή η συνεργασία ώστε να προχωρήσουμε σε πολιτικές απασχόλησεις που να είναι αποτελεσματικές. Κυρίως και διότι εν μέρη τουλάχιστον, εντάξει δεν νομίζω πως εδώ θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της ανεργίας, αλλά τουλάχιστον εν μέρη θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ε, στην ελάφρυνση του προβλήματος ε, για πολλούς. Εγώ θα ήθελα να σας πω τι ε, δράσεις ανέλαβα Καταρχήν προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε νέες ενδείξεις σε σχέση με αυτές που υπήρχαν. Ε, ζητήσαμε να εισαχθεί μια τροπολογία εντός της οποίας η αρμοδιότητα για τις εργασιακές πολιτικές να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έπειτα ε, έχουμε το Ρέντζι και το Job Act και όταν το ρωτάμε μας, ε, για αυτά τα θέματα κάπως μας φύγεται το στομάχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε πως ε, οι αρμοδιότητες για την απασχόληση θα πρέπει να παραμείνουν στα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσω είναι το γεγονός ότι στην Επιτροπή θα πρέπει να δοθούν εξουσίες για κατεξουσιδότηση πράξης και αυτό γιατί ε, αυτό αφαιρεί Μάλλον δεν θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα γιατί στερεί αυτό τη δυνατότητα συνεργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο, με εμά δηλαδή. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια τέτοια φάση δεν είναι αυτό απαραίτητο ούτε και σκόπιμο. Να πούμε δηλαδή ότι η πρόσβαση σε αυτές ε, τις βάσεις για τους ε, χρήστες να είναι επιπληρωμή Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολύ συχνά η μετακίνηση για να αναζήτηση εργασίας δεν είναι ε, κούσια, είναι αναγκαστική. Ε, ωστόσο εκεί η κινητικότητα, εκεί που είναι όντως επιλογή, καλό είναι να υπάρχουν τέτοια όργανα όπως το ΕΟΡΕΣ που διευκολύνουν την κατάσταση. Οι εθνικέ πολιτικές θα πρέπει να γίνουν βέβαια πιο αποτελεσματικέ, κυρίως όσον αφορά την εσωτερική απασχόληση. Και θα ήθελα επίσης, ε, και όταν θα κάνουμε τη συνάντηση των σκιωδών, θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ενταχθούν εδώ και αναφορές και όχι μόνο οικονομικοί δείκτες, αλλά και κοινωνικοί δείκτες, γιατί θεωρώ ότι συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές μεταβλητές, ενώ θα μπορούσε να είναι ένας καλός κανόνας που να θεσπίσουμε Τώρα, η πρόσβαση, και αυτό είναι θετική προστιθέμενη αξία, όταν δηλαδή επικοινωνούμε με αποτελεσματικό τρόπο και διευρυγμένο τρόπο για τις δυνατότητες που μπορεί να προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερο είναι αποτελεσματικές και μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει και να υποφεληθεί. Το χρησιμοποίησα και στην έκθεσή μου όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας Λέω λοιπόν στο συνάδελφο γιατί και εδώ να μην δημιουργηθεί μια, ένα application, μια εφαρμογή για τα smartphone ώστε να γίνεται πιο εύκολη η ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Δεν θα ήθελα αυτός, αυτή η μέθοδος της δικτύωσης στοιχείων και ευκαιριών να εξεταστεί με ελαφριά καρδιά γιατί οι νέοι έχουν μεγάλη άμεση επαφή ανάμεσά τους και ορισμένες ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφερθούν μέσω της Ευρώπης, ακριβώς μέσω τέτοιων ε, εργαλείων που είναι ε, ιδιαίτερα προσφυλή στους νέους, ε, να είναι θα είναι πιο αποτελεσματικά. Τη στιγμή που ένας εργαζόμενος πρέπει να ε, διαλέξει αν θα πρέπει να πάει σε μια άλλη χώρα για να δουλέψει, το έργο του ΕΟΡΕΣ δεν θα πρέπει να σταματά σε αυτό, αλλά να προβλέψουμε και πολιτικές ε, παρακολούθησης, στήριξης, ε, στήριξης για να δούμε πώς προχωρά στη νέα θέση επασχόλησης, στη νέα πραγματικότητα όπου θα ε, πρέπει να εργαστεί. Βοήθεια δηλαδή στήριξη στους εργαζόμενους. Όλα αυτά φυσικά δωρεάν. Συστήνουμε επίσης και μια ε, παρακολούθηση για τη διαφάνεια των ροών που θα πρέπει να δημοσιεύονται έτσι ώστε να δοθεί σημασία τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά. Κυρίως να προσπαθήσουμε να οθήσουμε την προσφορά, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολύ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενώ πολύ λιγότερη προσφορά και δεν προωθείται και επαρκώς. Ε, εντάξει, να ευνοήσουμε λοιπόν την απασχόληση γενικά. Επαναλαμβάνω την ε, πλήρη μου διάθεση για συνεργασία με τους συναδέλφους. Ε, δηλαδή το υποβάλλω πολλές τροπολογίες δεν σημαίνει επίκρισεις, όχι. Σημαίνει αναζήτηση καλύτερης και στενότερης συνεργασίας. Ευχαριστώ. Μαμ, the yours. <clears throat> Μαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν κανείς συντάσσει έκθεση και υπάρχουν 699 τροπολογίες, είναι μάλλον ε, ότι πρόκειται για μια κακή έκθεση. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν δείτε δε ε, τις τροπολογίες, θα δείτε ότι πολλές από αυτές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και είναι ενθαρρυντικό το στοιχείο αυτό. Το ερώτημα είναι, τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ε, αυτό που αποκαλείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη ε, αξία στο EURES. Ε, έχουμε και θετικά παραδείγματα όσον αφορά και τη συνεργασία και με γειτονικές χώρες. Και νομίζω ότι το δίκτυο EURES είναι ένα θετικό παράδειγμα. Γιατί όταν οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται, ε, αναζητούν εργασία, τότε χρειάζονται και τη βοήθεια των ε, θεσμικών οργάνων. Θέλουμε ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοποίηση των πόρων και θέλουμε να ε, επιτύχουμε το στόχο της εμβάθυνσης και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είπες ότι χρειάζεται εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Χάινς, αν, δεις την τροπολογία μου, θα δεις ότι θα πρέπει ε, οι κενές θέσεις να αποστέλλονται πρώτα στο γραφείο συντονισμού και υπάρχουν πολύ θετικέ εμπειρίες. Έχουμε στην Γερμανία για παράδειγμα τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ και αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει διάθεση συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και υπάρχει και απαραίτητη ποιότητα. Δηλαδή να μην, να μην ε, προσφέρονται απλά εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά να υπάρχει συνεργασία για να ε, υπάρχει και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα που αποτελεί αντικείμενο πολλών ε, τροπολογιών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μην δημοσιεύουν νέες, ε, κάποιες θέσεις εργασίας ανάλογα με, ορισμένες, ε, ε, με ορισμένα προσόντα. Για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία θέλω και θεωρώ σημαντικό να αποφύγουμε το φαινόμενο να αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης ε, ως ε, εύκολο τρόπο ε, προσκόμιση κερδών. Θα πρέπει να έχουν άλλο χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει άλλο χαρακτήρα η πρακτική άσκηση. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πολύγλωσσες δημοσιεύσεις θέσεων εργασία, Θα πρέπει να εξασφαλιστεί δηλαδή η πολυγλωσία, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι καθένας θα αναζητεί θέση εργασίας στην χώρα καταγωγής του. Χρειαζόμαστε δηλαδή καλές δημοσιεύσεις στη βάση της εμπειρίας που έχουμε συλλέξει και νομίζω, Χάνς, μπορούμε να εντάξουμε και ένα τέτοιο πνεύμα στην έκθεση και είναι πάρα πολύ σημαντικό η ενίσχυση της κινητικότητας να μην προβλέπεται απλά σε ορισμένα έγγραφα, αλλά θα ε, υλοποιείται και στην πράξη, ώστε να αυξηθεί και ο βαθμός συμφωνίας των πολιτών για το ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστώ, ο κύριος Λένος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάιντ Πέκερ για την έκθεσή του. Συμφωνώ με τον Τόμας ε, οι τροπολογίες και ο αριθμός τους ε, δεν ε, συνάδουν με την ποιότητα της ε, έκθεσης. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε συμφωνία για το κείμενο αυτό. Τρία σημεία θα θέλω να θέσω που είναι πολύ σημαντικά για μένα. Πρώτον, αν θέλουμε όντως να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της διασυνοριακής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα κράτη-μέλη που γειτονεύουν να ε, συνεργάζονται πολύ περισσότερο, να τονίσουμε τη σημασία ενός τέτοιου δικτύου όπως το EURES σε διασυνοριακό επίπεδο, γιατί μερικές φορές νομίζω ότι σε αυτές ειδικά τις περιφέρειες αν θέλουμε να αυξήσουμε την απασχόληση και να καταπολεμήσουμε την ενεργεία, πρέπει να μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος ε, μια τέτοιου είδους περιφέρεια, όπου κάποιος πρέπει να περάσει τα σύνορα για να βρει δουλειά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το επιβάλλουμε αυτό, αυτή τη διασυνοριακή προοπτική σε αυτήν την πρόταση. Επίσης, η ένταξη των δημοσίων εταιριών έβρεσης εργασίας των ιδιωτικών γραφείων έβρεσης ε, εργασίας. Μερικά κράτη-μέλη δεν έχουν τέτοιου είδους ε, ε, εμπειρία. Ίσως θα έπρεπε να τα συμπεριλάβουμε στο δίκτυο του Eures γιατί μπορεί να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία. Τελευταίο σημείο από τη δική μου την εμπειρία από τη δική μου χώρα πολλοί κόσμος ε, αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει από το εξωτερικό και έχει δουλέψει εκεί. Έχουν, έχει κάποιο πρόβλημα με τις φορολογικές αρχές σε σχέση με τη διπλή φορολόγηση. Δεν είναι πάρα πολύ σαφές ποιος φόρος πρέπει να πληρωθεί που. Ίσως θα έπρεπε να δούμε τις διμερείς φορολογικές συμφωνίες που έχουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους εντός του δικτύου Eures. Αν ενημερώνεται κάποιος ε, εργαζόμενος που κάνει χρήση της κινητικότητας, παρακαλούμε ενημερώστε τον και για το φορολογικό κομμάτι. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μην απογοητεύεται κανείς και να μην έχει πρόβλημα μετά και να μην είναι αποτρεπτικό αυτό το στοιχείο για κάποιον που θέλει να πάει να δουλέψει εκτός της χώρας του. Αυτά για μένα για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπέικερ. Είναι εξαιρετικό το έργο που επιτέλεσε πραγματικά. Για όσα ακούστηκαν, θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Και εγώ προέρχομαι από χώρα του Νότου, είμαι από την Πορτογαλία. Και όταν μιλάμε για κινητικότητα και διασυνοριακή δυνατότητα έβρεσης εργασίας, αναφέρεται πολύ συχνά ότι θα πρέπει να ε, υποχρεώνονται οι νέοι άνθρωποι να βγουν στο εξωτερικό δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να αποφασίσει να εργαστεί στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στη χώρα τους. Και αυτό κατανοητό είναι. Και εμείς πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα έβρεσης εργασίας στο εξωτερικό στους νέους ανθρώπους. Η νεανική ενεργία... Ε, έχει εκτιναχθεί. Και θέλω να πω ότι είναι ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την καταπολέμηση της και ε, να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα των νέων να ψάξουν δουλειά ε, στο εξωτερικό. Συμφωνώ και με την Έλληνα όσον αφορά τα ζητήματα τα φορολογικά. Και κάτι ακόμη για την κινητικότητα. Ε, αναφέρομαι στα προσόντα. Υπάρχουν νέοι με πολλά προσόντα που θα ήθελαν να εργαστούν στο εξωτερικό, αλλά αντιμετωπίζουν ε, δυσκολία γιατί δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών τους, τις, τα προσόντα τους. Και εκεί θα πρέπει, και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε στο επιθυμητό ε, αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχτάν, Μαχτάν, ζητήσατε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για το ΕΡΕΣ, ΙΡΕΣ, εμείς, ε, ε, εμάς, εμείς έχουμε πολύ δυσαρεστή φύση. Άκουσαμε όλα αυτά που υπόθηκαν. Τώρα το να μπορεί ο καθένας να βρει, ε, ειδικά αν είναι νέος, ε, μια εργασία κάπου στην Ευρώπη, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένας ευσεβής πόθος. Όμως έχουμε ένα φόβο ότι τελικά ε, κινητοποιούνται ε, ε, εργαζόμενοι σε χώρες που έχουν καμηλότερους μισθούς ε, προς χώρες που έχουν υψηλότερους μισθούς, αλλά ήδη σε αυτές τις πιο πλούσιες, ας το πούμε, χώρες έχουν, υπάρχει ήδη υψηλό ποσοστό ανεργίας ε, και υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι με διπλώματα, με πτυχία ε, που πηγαίνουν σε χώρες που, είναι πολύ, που τους υποδέχονται πάρα πολύ καλά ε, που έχουν, έχουν πολύ ψηλότερους μισθούς. Δηλαδή φεύγουν από τη μία χώρα, δημιουργείται ένα πρόβλημα όμω στην άλλη χώρα στην οποία πάνε. Μπορεί να λύνεται το πρόβλημα στη μία χώρα, αλλά να δημιουργούμε πρόβλημα στην άλλη. Υπάρχουν χώρε που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ιδιωτικά ε, γραφεία, ε, όμω ποιες ε, είναι αυτές που δουλεύουν για μεγάλους ομίλους, για παράδειγμα στα δημόσια έργα ή στην ε, στον τομέα των ναυπηγείων. Τελικά αυτό που κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά μεγάλους ομίλους που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη εξαθλίωση και εκμεταλλεύονται κόσμο που στη δική τους χώρα θα είχαν ε, πολύ χαμηλότερο μισθό, ε, δίνοντάς τους, δίνοντάς τους μισθούς διπλούς από αυτούς που θα είχαν στη χώρα τους, αλλά παρόλα αυτά στη χώρα στην οποία πάνε ο μισθός εξακολουθεί να παραμένει χαμηλός αυτό πραγματικά έρχεται σε αντίθεση με την επιβολή, με την επιβολή που θέλουμε ενός κατώτατου μισθού. Τελικά όμως εσείς αυτό κάνετε και γι' αυτό εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου και θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαντέ. Ευχαριστώ πολύ και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Θα ήθελα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, και να ε, επικροτήσω την εργασία του εισηγητή, τον ενθουσιασμό του και την αποφασιστικότητά του για το θέμα. Θα ήθελα και εγώ να επιμείνω στην αναγκαιότητα του να ληφθεί υπόψη η πτυχή, η διασυνοριακή ε, η κινητικότητα μπορεί να θεωρείται μια ευκαιρία, αλλά μερικές φορές ε, η βίωση της εμπειρίας αυτής είναι όχι πολύ καλή. Η πραγματικότητα η διασυνοριακή είναι μερικές φορές μια κατάσταση κάπως ε, ενδιάμεση, η οποία δίνει κάποιες καλές ευκαιρίες, έχει πολλά πλέον εκτήματα και γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω, όπως είπε και ο εισηγητής μας άλλωστε, ότι αυτή η διασυνοριακή κινητικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ενθαρρύνουμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το εργαλείο EURES θα λάβει υπόψη αυτή τη διασυνοριακή πτυχή. Το θέμα βέβαια της γλώσσας τίθεται όταν υπάρχει γενική φύσεως κινητικότητα. Όλο και περισσότερο ισχύει αυτό για την διασυνοριακή κινητικότητα. Εγώ ως Ευρωβουλευτής θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε όλοι να θέλουμε να ενθαρρύνουμε την εκμάθηση γλωσσών, όμως ε, μέχρι να γενικευτεί αυτή η εκμάθηση γλωσσών πρέπει και στο Γιουρές να σκεφτούμε εργαλεία τα οποία θα, θα επιτρέπουν ε, την ύπαρξη της πληροφορίας σε διάφορες γλώσσες, όπως είπε και ο συνάδελφος Τόμας Μαν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η κυρία Μωρά Σαρτιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επικροτήσω την δουλειά του συναδέλφου Μπέκερ, ο οποίος πραγματικά υπερασπίστηκε τόσο πολύ καλά και αύξησε και το δυναμικό του Γιουρές ε, και όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που πήραν το λόγο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στο Γερές δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία ε, αμφιβολία και εκεί όλοι όσοι έχουν τέτοιου είδους αμφιβολίες ε, ουσιαστικά πάνε κόντρα στην ιστορία. Είναι πολύ απλός ο λόγος ότι η κινητικότητα των νέων ε, όταν τους διευκολύνει το γιουρές τους δίνει ένα επιπλέον, ε, μια επιπλέον δυνατότητα να ε, μπουν στην αγορά εργασίας και σε αυτή την πρώτη φάση όταν διευκολύνονται από το γιουρές υπάρχει μετά ένα δεύτερο στάδιο ότι η γεωγραφική κινητικότητα αναπτύσσει την επαγγελματική κινητικότητα και αυτό είναι ένας ένας ε, παράγοντας ε, αξιοσημείωτος για να παραμείνει κανείς στην αγορά εργασίας. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οποιαδήποτε αναδίπλωση είναι, είναι μια εντελώς παροχημένη αντίδραση και το ε, πρέπει να είναι ένα επιπλέον εργαλείο που θα επιτρέψει στους νέους να καταπολεμήσουν την ανεργία. Αφήστε τους νέους εκεί το να αφήσετε τους νέους ε, εκεί που μένουν είναι σαν να επιτείνει κανείς το κίνδυνο ε, να μπουν σε ε, ανεργία, να, να, να είναι άνεργοι, ενώ το γιουρές τους δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης απασχολησιμότητας και μάλιστα πιο βιώσιμης. Γι' αυτό νομίζω ότι η δική μας πολιτική ευθύνη, από οποιαδήποτε χώρα και αν προεχόμαστε και από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα, πρέπει, ε, είναι να υποστηρίξουμε την έκθεση του κυρίου Μπέκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τις επεφημίες. Μήπως θέλει ο κύριος Μπέκερ να πει ορισμένα πράγματα πριν συνεχίσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα το επόμενο μισάωρο. Όχι, αστείευομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και να επισέλθω σε ορισμένα θέματα. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως θέματα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και με τους σκιώδους αλλά και όταν το ξανασυζητήσουμε το θέμα εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, θεωρώ ότι το αίτημα να υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα για εργαζόμενους και για μαθητευόμενους είναι αδιαμφισβήτητα. αδιαμφισβήτη. Εκεί όπου υπάρχουν οι δυνατότητες για θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης θα πρέπει αυτές να αξιοποιούνται. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση όταν κάποιοι λένε ότι τα μέλη θα αντικατασταθούν από τα κέντρα συντονισμού. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν δείτε το σημερινό σύστημα, το σύστημα όπως έχει σήμερα, και λάβει υπόψη το γεγονός ότι το ποσοστό κινητικότητας στην Ευρώπη είναι 0,3% σχεδόν αμεληταίο δηλαδή, ενώ στη ΣΥΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20 φορές υψηλότερο, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να συζητούμε βελτιώσεις. Και νομίζω ότι είναι λογικό το να υποστηρίξουμε αυτήν την νέα ε, πλατφόρμα. Θα χρειαστούν βεβαίως και εκστρατείες ε, γνωστοποίησης, δημοσιοποίησης του νέου συστήματος, διότι δεν μπορεί ένα τέτοιο νέο σύστημα να είναι αποτελεσματικό αν οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν στον ε, κύκλο των ε, γνωστών μου δεν το ήξερε σχεδόν κανείς το σύστημα. Μπορεί να φταίνει και οι φίλοι μου, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά είναι ενδεικτικό. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται και η άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρίες και στο ίντερνετ. Άρα, συνεργασία και συντονισμός θα πρέπει να υπάρχει σε αυτήν την δεξαμενή κενών θέσεων ε, εργασίας. Και δεν θα πρέπει να υπάρξει, δεν θα πρέπει να προβλέπεται προτιμησιακή μεταχείριση για ορισμένες εθνικές θέσεις εργασίας. Αυτό δεν θα ήταν ευρωπαϊκή, δεν θα, δεν θα, δεν θα εξασφάλιζε την ευρωπαϊκή διάσταση και να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει χρέωση για όσους αναζητούν εργασία και θα πρέπει αυτό να το εξασφαλίσουμε. Για τις διασυνοριακές συνεργασίες νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Είναι ένα από τα στοιχεία ε, με ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρα. Για τους ελέγχους. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν και προβλέπονται. Για την ε, εμπλοκή και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Να απαντήσω στον Τόμας Μαν Μα είναι προφανές ότι η σημασία των κοινωνικών εταίρων είναι αυτονόητη, ιδιαίτερα στα ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, που αλλού άλλωστε. Και νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε και σε αυτό το σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ποιοτική κινητικότητα. Ναι, συμφωνώ. Δεν θέλουμε να ε, έχουμε στόχο το dumping προφανώς. Θα πρέπει να μιλούμε για θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Επίσης, δεν θέλουμε το Γιούρες να είναι μια απλή στοσελίδα, αλλά ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής για την αγορά εργασίας. Επίσης μου άρεσε αυτή η ε, αναφορά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Νομίζω ότι θα πρέπει και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου να εξετάζεται πόσο και ε, σε ποιο βαθμό το κάθε κράτος μέλος αξιοποιεί αυτό το δίκτυο τόσο για την αγορά εργασίας όσο και η, βεβαίως η, εθνική εργασ, αγορά εργασίας και τα μέτρα στήριξης αποτελούν και εξακολουθούν να αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και συγκεκριμένε ε, υποχρεώσεις από την πλευρά των κρατών μελών. Κατάργηση των διακρίσεων. Συμφωνώ και σε αυτό. Συνάδελφοι, ε, τα σχόλιά σας ποτέ δεν τα εκλαμβάνω ως ε, επικρίσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την αυταπάτη ότι το Γιούρες θα μπορέσει να εξαλείψει πλήρως την ε, ανεργία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο το Γιούρες. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ε, ενισχύσει ή να ε, επιταχύνει ορισμένα μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας. Διότι αν τα κρατη συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να αναλάβουν δράση, αυτό είναι σημαντικό και θα μπορέσει να υπηρετηθεί ο στόχος αυτός και μέσω του Ιούρες. Κοινωνικοί δείκτες. Το ποιοι θα πρέπει να είναι αυτοί θα το εξετάσουμε, αλλά είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα το συγκεκριμένο. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, για εφαρμογές, smartphone κτλ. κτλ. Αλλά σε πρώτη φάση βεβαίως πρέπει να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του συστήματος στον υπολογιστή. Για την προστασία των όσων ε, φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, συμφωνώ. Ε, όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ορισμένους ε, δημοσιονομικούς περιορισμούς. Και φτάνω στις ε, τελικές μου παρατηρήσεις. βεβαίω, δεν θα πρέπει να υπάρξει κατάχρηση των θέσεων πρακτικής εργασίας και μαθητείας, ούτε να ε, αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την εξέβριση φθηνού εργατικού δυναμικού. Εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε τον σεβασμό που ε, τρέφουμε και την υποστήριξή μας στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των νέων ανθρώπων. Πολυγλωσία, πολύγλωσσες ε, δημοσιεύσεις, συμφωνώ απόλυτα και με αυτό. Βεβαίως όλες αυτές οι αρχές δεν θα πρέπει απλώς να ε, καταγράφονται στα χαρτιά, αλλά ξαναλέω ότι όταν η κινητικότητα κινείται στα επίπεδα του 0,3% υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, βελ... περιθώρια βελτίωσης για τις ε, ανάγκες, την εξυπηρέτηση, τη στοχευμένη εξυπηρέτηση αναγκών των περιφερειών, θεωρώ ότι και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας αποτελούν ήδη ε, συστατικό στοιχείο αυτού του έργου και όσον αφορά προβλήματα φορολογικής φύσης ή προβλήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση θα τα εξετάσουμε και αυτά. Οι νέοι άνθρωποι, βεβαίως κυρία Ρομπέρο, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να φύγουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Αυτό θα ήταν η απόλυτη παρανόηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των νέων ανθρώπων. Τίτλοι σπουδών και προσόντα. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των προσόντων. Νομίζω ότι το η ύπαρξη του Γιούρες θα αναγκάσει σε ένα βαθμό τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα πράγματα και στον τομέα της αναγνώρισης των προσόντων νομίζω ότι η κινητικότητα από χώρε χαμηλού εισοδήματο σε χώρε υψηλότερου εισοδήματο είναι πρόβλημα. Διότι αν κάποιο ε, κράτος κράτο μέλο υψηλού εισοδήματο έχει κενέ θέσει εργασία, τότε θα πρέπει να μπορεί να ε, αναζητεί ε, ανθρώπους για την κάλυψη των θέσεων αυτών σε όλη την Ευρώπη. υπάρχουν συγκεκριμένες ε, νομικές διατάξεις για τις αμοιβέ σε κάθε κράτος μέλος και ε, άρα από αυτή την άποψη ε, δεν υπάρχει κίνδυνος. Επίσης, θεωρώ ότι η συνολική προσέγγιση της Κομισιόν είναι θετικό, θετική. Και κύριε Σαντιένε, ναι, έχετε δίκιο. δεν πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω το, οι δυνατότητες του Γιούρες είναι εξαιρετικά υψηλές. Και αυτή η παροχή της δυνατότητας έβρεσης εργασία για του νέου ανθρώπους νομίζω ότι είναι το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Ε, χαίρομαι για τη συνεργασία με όλους τους ε, σκιώδει και είμαι βέβαιος ότι τι επόμενε εβδομάδε θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ, ευχαριστώ για όλους τους ομιλητέ για τι παρεμβάσει του και τα σχόλιά του. Θα ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Ριμπέρη και στην κυρία Σαντιέ, αλλά να σας δώσω κάποιες πληροφορίε για το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Ε, έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, αυτής της έκθεσης για το Γιούρες θα γίνει στις, η ψηφοφορία θα γίνει στις 7 Μαΐου. Υπάρχει ένα, μια αλλαγή δηλαδή στο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, Για το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα μπορέσουμε σήμερα, δεν θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε σήμερα. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η ε, Μαρτίου και η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει στις 24 Μαρτίου. Μιλώ για την απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής ε, Κοινωνικής Προστασίας και την κατάρριξη της απόφασης. Υπάρχει επίσης ε, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 3 Μαρτίου και έγκριση στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου. Για το 15 τη σημερινή διάταξη την αστική διάσταση στι πολιτικέ τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ανέφερα, η Ευελίν Ρέγνερ δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα, αλλά μου έχει δώσει κάποιες σημειώσεις της και λέει η κυρία Ρέγνερ ότι το σχέδιο γνωμοδότησης θα επικεντρώνεται σε πέντε σημεία. Πρώτον, οι Δήμοι και οι πόλεις θα πρέπει να ε, εμπλέκονται στη διαδικασία. Δεύτερον, οι περιφέρειες θα πρέπει να εμπλέκονται στο πρόγραμμα επενδύσεων. Θα πρέπει τρίτον να υπάρχουν ε, επενδύσεις και δεν θα πρέπει να ε, συνυπολογίζονται στο δημόσιο χρέας. Επίσης, θα υπάρχει μια διάσταση για τα φύλλα, για την ισότητα των φύλων Και πέμπτον, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Και όσον αφορά το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, θα υπάρχει δυνατότητα, ε, θα, σα σας δώσω τη δυνατότητα και θα, να κάνετε παρεμβάσεις. Θα ήθελε η ίδια να τονίσει ότι οι πόλεις και οι δήμοι ε, αποτελούν καθοριστική σημασία παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και αναμένει τις τροπολογίες όλων σας και τη συνεργασία βεβαίως με τους σκιώδεις τις Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η Μαρτίου και η έγκριση στην Επιτροπή θα γίνει την 1η Απριλίου. Επιστρέφουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Πολύ σημαντική έκθεση και αυτή για τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και για μας εδώ στην Επιτροπή μας. Και δίνω το λόγο στην κυρία Μογάν Σαρτιέ. Merci, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ε, τους ναυτικούς που τροποποιεί κάποιες οδηγίες που ήδη υφίστανται. Γιατί, γιατί στην ε, ενωσιακή νομοθεσία οι ναυτικοί, θα σας υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό, αποκλείονται από κάποιες οδηγίες που οργανώνουν την προστασία των εργαζομένων. Επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά όλοι μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιωδών εισηγητών, ε, την Ανιές, ε, την Ούλα, από τους φιλελεύθερους ε, και από τους σοσιαλδημοκράτες, τον Πατρίκ από την ΚΟΕ, την Τζίν από τους Πράσινους και την Κέισια για τους ελεύθερους δημοκράτες που πραγματικά συνεισέφεραν πάρα πολύ στη δουλειά μας για στρατηγικούς λόγους ε, και βασίστηκα πάρα πολύ στην ε, γραμματεία της Επιτροπής μας, ε, θα θέλησα να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες όλες από την αρχή της δουλειάς μας και γι' αυτό το λόγο κάναμε μία συνάντηση εισηγητών μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και με τους εκπροσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για το θέμα μας. Μετά λοιπόν το σχέδιο έκθεσης ε, Κατατέθηκαν 34 τροπολογίε, 2 από το ΕΛΚ, 19 από του Σοσιαλδημοκράτε, 2 από την ECR, 2 από του Φιλελεύθερου, 1 από του πράσινου και 5 από του ελεύθερου δημοκράτε και 3 από του μη εγγεγραμμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που συνεισέφεραν με πολύ επικοδομητικέ τροπολογίες και που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της, ε, του συνόλου της δουλειάς ε, που αποκρισταλώθηκε σε αυτή την έκθεση και ε, χαίρομαι πολύ που μεταξύ των τροπολογιών αυτών 16 από τις 34 είναι σχεδόν ταυτόσιμες με αυτά που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην έκθεση προσπαθήσαμε να ε, ενσωματώσουμε και να συγκεράσουμε τις διάφορες απόψεις και νομίζω ότι αυτό ε, θα είναι εύκολο. Η ιδέα των περισσότερων ε, εισηγητών είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των πλειοκτητών. Εκτός από αυτές τις 16 ταυτόσιμε τροπολογίε. κάποιες τροπολογίες είναι απολύτως συμβατέ με την έκθεση από τη μία και από την άλλη με την συμφωνία που προανέφερα και αναφέρομαι κυρίως στην τροπολογία 19 του Ζερόμ Λαβριγιό που τονίζει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην περιεκτική ανάπτυξη, όπως επίσης και τροπολογία 22, ε, των σοσιαλδημοκρατών ε, για τη σημασία της σύμβασης ε, της, της εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας για την συνθήκη, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην ναυτιλία. Τροπολογία 21 και 23 Μα ζητούν προσοχή για το φόρτο εργασίας ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Και βεβαίω ε, πολλοί επανεπισημαίνουν τη σημασία της βελτίωση των συνθήκων εργαζομένων των ναυτικών αυτό είναι ο γενικό μα στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τζιν που φεύγει τώρα αλλά που πραγματικά είσαι πολύ δραστήρια στο θέμα αυτό τα προβλήματα τα τεχνικά που μπορεί να ε, παρουσιαστούν ε, θα τα επιλύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιβεβαιώνοντας ε, τι μπορεί να, να... συμπεριληφθεί. Κάτι τεχνικό λοιπόν που θα ήθελα να πω για την τροπολογία 18... Είμαστε σε μία νομοθετική έκθεση και σε αυτή την νομοθετική έκθεση δεν μπορούμε να αναφερόμαστε παρά μόνο σε υπάρχοντα επίσημα κείμενα. Σήμερα λοιπόν η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των πλειοκτήτων δεν είναι ένα επίσημο κείμενο. Επομένως μπορούμε εμείς να το συμπεριλάβουμε στον προβληματισμό μας και στις εργασίες μας αλλά δεν μπορούμε να παραπέμπουμε σε αυτό ε, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία της εργασίας μας ε, για τις τροπολογίες σε σχέση με τη συμφωνία που μόλις προανέφερα, στην έκθεσή μου θα θυμάστε ότι εισήγαγα την αναφορά στις νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ε, ε, ενσωμάτωση της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων. Είναι ένα σημείο επί του οποίου όλες οι πολιτικές ομάδες, ε, οι περισσότερες ε, συμφώνησαν, κάποιες άλλες ομάδες είναι κάπως πιο επιφυλακτικές. Ε, κοιτάξτε, θα έχουμε μία ακόμη συνάντηση που θα γίνει στο Στρασβούργο στις 12 Μαρτίου κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες ε, όσο το δυνατόν πιο ευρείας συνένεσης και θα λάβουμε υπόψη και την άποψη της Επιτροπής Αλείας ε, η Βερόνικα Λοπέ Φοντάνιε ε, συνεισφέρει τα μάλα. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες με την Επιτροπή Αλίας. Και θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω κάποιες, κάποια γλωσσικά σφάλματα μεταξύ της δικής μου έκθεσης που ήταν στα γαλλικά και της αγγλικής ε, εκδοχής. Θα ήθελα να πω ότι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 η τροπολογία 15 για την αναφορά στην παράγραφο 1 και 2. 1 και 2 κάτι το οποίο θα προσθεθεί για να είμαστε σύμφωνοι με τους κοινωνικούς εταίρους και το ε, ίδιο το transferer θα γίνει transferir για να είμαστε, από, να, είμαστε να συμφωνούμε με, την, ε, με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτά ήθελα λοιπόν να σας πω. Θα ήθελα τώρα να ακούσω τις απόψεις των ε, διαφόρων ε, σκιωδών εισηγητών για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει ο χρόνος μας. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω τους σκιώδες να ε, είναι πολύ ακριβείς και σύντομοι. Η ε, κυρία Γιονκέρης από το Σοσιαλιστή. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και για τη δουλειά που κάνατε. Να σας πω το εξής. Ε, η ομάδα του ΕΛΚΑ, του, των Σοσιαλιστών, με συγχωρείτε, στηρίζει τις βασικές γραμμές της έκθεσής σας ακριβώς λόγω του ότι στηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και ε, προσπαθεί ε, να δουλέψει ε, με αυτή την έκθεση. Είναι καλό που γίνεται αυτή η συνεδρίαση γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι είμαστε σε θέση να εργαστούμε και να επεξεργαστούμε τα, τις τροπολογίες που αφορούν κυρίως τα εκτιμώντας Όντως ε, βελτιώνεται η κατάσταση για τους ναυτικούς, ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τη σύγχρονη τεχνολογία. Ε, που βελτιώνει την ζωή των ε, ε, ναυτικών εφόσον υπάρχουν γιατί να μην τη χρησιμοποιείς. Αυτή είναι η δική μου συμβολή. Είμαι πεπισμένη ότι θα συνεργαστούμε θετικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. I give the floor to Mr. Gericke from ECR. Ευχαριστώ, κύριος Γκερίκη από το ECR. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική τη συνεργασία. Νομίζω πως έχουμε φτάσει σε μια καλή έκθεση. Καταρχήν, λάβαμε υπόψη τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους Εγώ Ε, πρότεινα μόνο να αναφερθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δύο διαφορετικά σημεία γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη θέση των μικρομεσαίων στην οικονομία αλλά πρέπει να μείνουμε ανταγωνιστικοί να μην χάσουμε απέναντι σε φτηνότερες χώρες αυτό δεν είναι λύση Ωστόσο, οι δικαιότερες συνθήκες θα πρέπει να ισχύσουν για όλους και αυτή είναι η τροπολογία 21. Στη δεύτερη τροπολογία μου αναφέρομαι στο κόστος που προκύπτει από τις αλλαγές για τις μικρές εταιρείες. Και γι' αυτό το λόγο κάνω έκκληση να επικεντρωθούμε στα νομικά ζητήματα και να εξασφαλίσουμε την ε, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, διότι είναι σαφές ότι ο λόγος για τον οποίο εξετάζουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον θαλάσσιο τομέα και η προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντλαμπάγιοβα από τους Άλντε. Μιλώ εκ μέρους της Ούλα Βουτνάης. Θα ήθελε η Ούλα να ευχαριστήσει για την καλή συνεργασία και τις τροπολογίες των, ε, αυτού του θέματος. υπάρχει συμφωνία των κοινών εταίρων που πρέπει να ε, γίνει σεβαστή. Καταλαβαίνω από το ζήτημα για το οποίο έθεσα τροπολογία ήταν ε, γλωσσικού χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν έλθει σε συμφωνία, οι ομάδες ε, υπέβαλαν τροπολογίες που αποκλίνουν από αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συμφωνία που, στην οποία κατέληξαν ε, οι κοινωνικοί εταίροι είναι, χαρακτηρίζεται από ευαισθητία, θεωρώ ότι αυτό είναι ατυχές. Οι συμφωνίε των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ και όχι να αλλάζουν από τους ε, πολιτικούς φορές. Οπότε, εκ μέρου της Ούλα, θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή και τις σκιώδους και να εκφράσω ε, την ε, ικανοποίησή της και την προθυμία της για περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Γέρικα από την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μογέν Σαχτιέ για τη δουλειά της. Οι ναυτικοί είναι άνθρωποι που δουλεύουν πολύ σκληρά. Σε κάθε κατάσταση σε κάθε θαλάσσια συνθήκη, δηλαδή πολλές φορές ε, ε, κινδυνεύουν και γι' αυτό ήταν ανομαλία το ότι δεν περιλαμβάνονταν στο κοινοτικό κοινωνικό δίκαιο. Αυτό ήταν μια ανομαλία και έπρεπε γι' αυτό να διορθωθεί. και να προτείνει έτσι την ε, συμφωνία ε, που θα συζητείται με βάση το δίκαιο ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια σειρά πολύ θετικών ε, τροπολογιών. θα εξαρτηθεί από μας να το υιοθετήσουμε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα τον έφερα αυτό. 1η ε, Απριλίου ε, θα πρέπει εμείς να το εγκρίνουμε και η πρώτη Ολομέλεια του Μαΐου θα περάσει από την Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Να πω γεια σας και καλωσορίσατε σε όλους τους νέους που επισκέπτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν θα, Δεν θα συνεχίσουμε για πάρα πολύ ώρα, αλλά ελπίζω κάτι ενδιαφέρον να βρείτε, να ακούσετε στη διάρκεια της επίσκεψής σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τη Διεθνή Σύμβαση για τα... Ε, μάλλον τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης Εκδοση πιστοποιητικών και τήρηση φυλακών για το προσωπικό των αλληλευτικών σκαφών. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία στη βοήθεια που μου προσέφερε στην επεξεργασία αυτή τη έκθεση. Ήταν πολύτιμη. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διορθάσουν ε, τα, τις, τα, τις διατάξεις με βάση τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα αλληλευτικά σκάφη. Αυτή η σύμβαση υιοθετήθηκε το 1995 και ε, την έχουν ε, επικυρώσει 22 κράτα-μέλη. Μόλις τέσσερα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή και στόχο έχει να εγγυηθεί ότι το προσωπικό ε, στα σκάφη, στα ληφτικά σκάφη, θα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εργασία αυτή και την κατάλληλη ε, κατάρτιση επίσης. Ε, θα πρέπει αυτά να επιβεβαιώνονται μέσω επίσημης πιστοποίησης. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια επαγγελματική κατάρτιση που μετά αυτή βοηθάει στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, να κυρώσει αυτή τη σύμβαση εάν τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν, να... δεν την κυρώσουν. Όμω ούτε τα κράτη-μέλη μπορούν να την κυρώσουν διότι δεν έχουν άμεση ευθύνη, ε, αρμοδιότητα αν δεν του δοθεί η άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχει κανείς την ε, ε, κατάλληλη έγκριση από το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο ώστε να μπορέσουν να πικυρώσουν, να κυρώσουν. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη σύμβαση παρά μόνο τέσσερα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουν να κράτη-μέλη να κυρώσουν μια τέτοια σύμβαση που στόχο έχει να ευνοήσει την επαγγελματική κατάρτιση και να μειωθούν κατά αυτόν τον τρόπο και τα ατυχήματα. Μια πρότασή μου είναι λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να ε, υπερψηφίσει αυτήν την πρόταση του Συμβουλίου. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ε, ήρθα σε επαφή με τους κοιόδες συζητητές και ζήτησε τα σχόλιά τους ώστε να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε την έκθεση αυτή. Και χάρη στη συμβολή των συναδέλφων, δηλαδή ε, από την ΚΟΣΕΚΑ, την ΓΟΠΑ ΚΟΣΕΚΑ, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, θα πρέπει να είναι αυτή η έκθεση πέρα από την κινητικότητα, πέρα από την κατάρτιση. Ε, εδώ αυτό που διακυβεύεται είναι η ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασία. Ε, πρόκειται για συλληφτικά σκάφη συγκεκριμένων διαστάσεων. Δεν είναι παγκοσμιοποιημένε οι προδιαγραφέ και θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβουλέψει την Κομισιόν και το ε, Συμβούλιο να λάβουν αποφάσει σε σχέση με τους όρους κατάρτισης των ναυτικών και των αλλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρμονίζοντας τις διαδικασίες κατάρτισή τους, ε, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η αλληλεία είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα που, γνωρί... που συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα Έχουμε χιλιάδες κόσμο ωστόσο που δουλεύει πάνω στα λευτικά σκάφη και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από το Ευρωκοινοβούλιο να ε, προτείνει να ε, εγκριθούν, ε, μάλλον να κυρωθεί αυτή η σύμβαση, ώστε οι αλληλείς μας να είναι καλύτεροι στη δουλειά τους και να δουλεύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για να σχολιάσουν. Yes, well, uh, the floor is open. Ωραία, ανοίγει ο κατάλογος ομιλητών. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Ντλαμπάγιοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και πάλι, εκπροσωπώ την Ουλα Τούρνες. Μιλώ εκ μέρους της, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για όλους του τους εκθέσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να πει ότι το υποστηρίζει πλήρως. Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία τον τελευταίο Νοέμβριο για το θέμα αυτό. Και θεωρούμε ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων σε όλες μας τις εργασίες. Θα ήθελε η Ούλα επίσης να, αξιοποιήσει την ευκαιρία και να υπενθυμίσει την συζήτηση που έγινε στις 26, το 26 Νοεμβρίου που έγινε μεταξύ των εργοδοτών και εργαζομένων και τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν οι εταίροι. Είναι σημαντικό να ε, τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τα ζητήματα απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ούλα λοιπόν χαίρεται για το έργο που θα γίνει στο θέμα αυτό. Η κυρία Τζέντιλε έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς ημερίζομαι πολλές από τις ε, αναφορές ε, της εισηγητρίας. Νομίζω πως είναι όλα αυτά χρήσιμα για να δούμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά ε, στη θάλασσα ε, και άρα πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν οι ναυτικοί, να δουλεύουν με ασφάλεια και κυρίως μέσω ε, τέτοιων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης που να είναι πραγματικά χρήσιμα. Έτσι ώστε δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος προσοχής προς ένα κομμάτι της οικονομίας που ίσως τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της ε, Νότιας Ευρώπης, ε, έχει υποστεί για άλλους λόγους, για άλλα... Ε, λόγω άλλων επιλογές, έχει επιβραδυνθεί η θάλασσα μπορεί να είναι μια τεράστια ευκαιρία για να δημιουργηθούν ε, ε, καλές ευκαιρίες για εργασία και η θάλασσα μπορεί να αποτελέσει μια εξαίρετη ευκαιρία για ανάπτυξη αν όμως καταφέρουμε να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει κάτι τέτοιο, η εργασία, η ποιοτική εργασία περνά μέσα από την κατάρτιση κυρίως για το θέμα της ασφάλειας. Έχω την ε, εντύπωση ότι αυτή η ε, Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την ταχεία έγκριση αυτού του, αυτής της έκθεσης, διότι έτσι ο, ο κόσμος της εργασίας αλλά και οι ε, αλλιευτικές ε, εκμεταλλεύσεις περιμένουν ε, με ανυπομονησία τα πορίσματά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρικε. Όχι, δεν θέλεις να πεις κάτι για το ΙΣΙΑΡ. Ε, ήσουν στο δικό μας κατάλογο ως ε, σκιώδης, αλλά τότε πάμε στην κυρία Ζουμπέρ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς εν γέννη συμφωνούμε με τα όσα προτείνονται στην έκθεση. Στην ουσία πρόκειται για συγκατάθεση προς μια σύσταση του Συμβουλίου, οπότε δεν χρειάζεται ε, να μιλήσω επί γιατί συμφωνούμε με μια τέτοια απόφαση. Έχουμε την ε, εντύπωση όντως ότι αυτή και η οκύρωση μάλλον αυτής της σύμβασης από πλευράς των κρατών μελών θα βοηθήσει στην βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και άρα στην βελτίωση της ε, ασφάλειας των ναυτικών και των αλλιέων. Ε, εν τω μεταξύ, όμως τίθεται και ένα θέμα στην αιτιολογική έκθεση ε, που νομίζω πως είναι ενδιαφέρον και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η ε, Επιτροπή καλύπτει μικρά μέχρι μεσαία σκάφη. Ωστόσο θα πρέπει να, έχουμε να γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της αλίας, της, βιομηχαν... της, της μικρής αλίας και της βιοτεχνικής αλίας δεν καλύπτονται από τους κανόνες που θεσπίζει αυτή η σύμβαση. Ακριβώς αυτή όμως η αλληλεία είναι που είναι πιο ευάλωτη, πιο αβέβαιη και όπου η δουλειά τους και τα ωράρια εργασίας τους είναι λιγότερο ρυθμισμένα και σήμερα Εκ των πραγμάτων η απόδοση αυτών των εργαζομένων είναι πολύ χαμηλή και υπάρχουν και συμβαίνουν ατυχήματα που πολύ συχνά είναι θανατηφόρα και που, όπως μου εξήγησαν πολλές φορές, έχουν να κάνουν ε, με έναν απίστευτο αριθμό ορών στη διάρκεια των οποίων εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαρτήσουμε τούτη την προστασία μάλλον αυτών των εργαζομένων από την σύμβαση μόνο. Θα πρέπει να υπάρξει και κοινοτική νομοθεσία ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν εγγυημένο μίνιμουμ εισόδημα και ε, ε, μίνιμουμ ε, όρους εργασίας. Ε, πολλές φορές ε, τρέχουν και ακραίους κινδύνους. Τουλάχιστον στη χώρα μας, στην Πορτογαλία, ε, πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα και είναι κάτι που είναι απαράδεκτο. Thank you all for staying. Ευχαριστώ όλους όσοι έμειναν και που υπέβαλαν τα σχόλιά τους. να σας ενημερώσω για το, για το χρονοδιάγραμμα. Έγκριση στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει 24 Μαρτίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου. Σας ευχαριστώ όλους για την συμβολή σας και τη συμμετοχή στη συζήτηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ξαναξεκινούμε στις 3 το απόγευμα. Θα υπάρξει ακρόαση, την οποία συνδιοργανώνουμε με την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Ακρόαση για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη ως τρόπο για να καταμπολεμηθεί η ανεργία των νέων και η πρόρη εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εξετάζουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να βρεθείτε εδώ, να συμμετάσχετε, να ακούσετε και τους νέους ανθρώπους που θα μας μιλήσουν, αλλά να ακούσετε και εκείνους που ε, εργάζονται σε στενή συνεργασία με αυτούς τους νέους ανθρώπους. Οπότε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στις 3.